Καλησπέρα, συνάδελφοι. Θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Ζητώ συγγνώμη που χρειάστηκε να προβλέψουμε σε 9 τη νύχτα συνεδρίαση, αλλά δεν είχαμε δυνατότητα να οργανώσουμε άλλη τη συνεδρίαση. Θα εγκρίνουμε την ημέρα διάταξη εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Και δεύτερο σημείο τη ημερήσια διάταξη, τι ανακοινώσει του Προέδρου για τι συστάσει των συντονιστών, να πω ότι στη συνάντηση τη 15η Μαου οι συντονιστέ αποφάσισαν να ακυρώσουν την αρχικώ προβλεπόμενη αποστολή στη Ρουμανία να οργανώσουμε ανταλλαγή απόψεων με το Ίδρυμα για την Ανοιχτή Κοινωνία και την κατάσταση των ε, γυναικών ε, μουσουλμανικής θρησκείας στην Ευρώπη, να συντάξουμε προφορική ερώτηση για τα δικαιώματα των γυναικών στα Δυτικά Βαλκάνια και για γνωμοδότηση το 2019 να την αναθέσουμε στους σοσιαλιστές και δημοκράτες του χρόνου να οργανώσουμε στην ε, Παγκόσμια Μέρα για τις Γυναίκες ε, κάτι, κάποια εκδήλωση για τη συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψη πολιτικών αποφάσεων. Σημείο 2.2. Καλωσορίζουμε νέα μέλη στην Επιτροπή Γυναικών. Καλωσορίζουμε τον κύριο Ζωζέ Ιγνάσιου Φαρία από το ΕΛΚ. Καλώ ήρθατε στην Επιτροπή μας ως αναπληρωτής. Και Περνάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έχουμε να ψηφίσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ισορροπία επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Έκθεση της κυρίας Κοσλόφσκα Ράγεβιτς. Γνωμοδότηση μάλλον της κυρίας Κοσλόφσκα Ράγεβιτς και ξεκινάμε να ψηφίζουμε ευθύ αμέσω. Είστε έτοιμοι συνάδελφοι. Έχετε τις κάρτες σας. Α, ξεχάσατε την κάρτα σας. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε σε κάποιον. Yes, we will start. we will start. Να ξεκινήσουμε. Τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ποια?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 Συμβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 327. Όχι, 326. 326 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θέλετε να κάνουμε έλεγχο. Ωραία. Ήταν σαφές, αλλά Ας ξαναψηφίσουμε διανάταση ισχυρός υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 325 υπέρ. Κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά καλύτερα να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 272-273 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Έλεγχος. 272-273. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. 16 υπέρ κατά αποχές να κάνουμε έλεγχο για τη 16 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 334 υπέρ κατά αποχές έλεγχος 334 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. 333 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ωραία, έλεγχο. 333 ελέγχουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 32. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 33. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 34. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 35. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 36. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 375. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 376. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 377. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 378 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 157 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 37 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 38 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 39 υπέρ. 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πρέπει να κάνουμε έλεγχο. Για την, ε, συγγνώμη, τριοπολογία 21, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 3,99 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 400 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τέσσερα με προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 422, 422 υπέρ, κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε 422, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, απορρίπτεται. 423 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβεβαστική 41 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θέλετε να κάνουμε έλεγχο για την τροπολογία 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 456-457 καταπίπτουν 430 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 434 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 435-437 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 440 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 442 υπέρ κατά αποχές πρέπει να κάνουμε έλεγχο για την 442 442 άρχεται ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. ...443 υπέρ, κατά αποχές πρέπει να κάνουμε έλεγχο για την 443 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 έλεγχος άρχεται η φοφορία. πέρας απορρίπτεται 445 445 υπέρ κατά αποχές πρέπει να κάνουμε έλεγχο. 445 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 444 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εντάξει λοιπόν, έλεγχος 26, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 447 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 448 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 42 και 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για την 28 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. 454 υπέρ, κατά, αποχές, πρέπει να ελέγξουμε. 454, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, εγκρίνεται. Συμβεβαστική 44 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 468 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Πέρας εγκρίνεται. 471 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 472 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική πρώτη 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 38 υπέρ κατά αποχές έλεγχος έλεγχος για τα 38 άρχεται ψηφοφορία πέρας Απορρίπτεται. 39 και 40 ταυτόσημες υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά Ναι, με συγχωρείτε, έχει πάει 10. 58 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Για την 65. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 98 υπέρ. Α, καταπιεπτή. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 95. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να κάνουμε έλεγχο για την 95. Άρχεται ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 96. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Ναι, 10. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 13 συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 156 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε 156 Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 170. 170 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 183. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θέλετε έλεγχο 189 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Πέρα, ε, απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 190 υπέρ. Κατά. Αποχές. 190. 190 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 194 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 197 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Έλεγχος για την 198. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 199 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε για την 199. Πέρας. Απορρίπτεται. 202, 202 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 200 υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 201 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 204 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 205 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε τη 205 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 206 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 211 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Now the final word, Which one? Συνάδελφοι, να πάω στη σελίδα 26 πάλι. Τετρακόσια 27 για τους S&D. Σελίδα. Μετά την τροπολογία 24. 456 και 457 μαζί. 456-457 υπέρ. Κατά. να κάνουμε έλεγχο. 456-457. Απορρίπτονται. Και επόμενη 4-2-7. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Και τώρα τελική ψηφοφορία. Σχέδιο γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. τολ thank you very Να ευχαριστήσω και τους σκιώδες εισηγητές. Αυτή είναι η θέση μας. Ε, ε, πρέπει να εργαστούμε σκληρά στο εξής. Ε, Επόμενη συναδρίαση 20 Ιουνίου στις 9. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Τα λέμε αύριο. Good night. Καλό βράδυ σε όλους.